Κυρίες και κύριοι, αυτή η αίθουσα δεν παρέχει τις ευκολίες ενός καφέ, δεν είναι εστιατόριο, άρα αν θέλετε να πάρετε ένα αναψυκτικό, να δροσιστείτε, τέλος πάντων παρακαλώ να βγείτε και όσοι έχουν ακόμη κουράγιο να εργαστούν, να παραμείνουν, γιατί έχουμε πολλά θέματα ακόμα. Μάλλον δεν πίστηκαν όλοι, θα πρέπει να επιμείνω. Ε. Να περάσουμε λοιπόν τώρα, αν συμφωνείτε, στο επόμενο θέμα της μερίσιας διάταξης, δηλαδή περιουσιακές σχέσεις και καταχωρημένους, ε, περιουσιακές σχέσεις και καταχωρημένων συντρόφων. Είμαι συγκεκριτής και για τις δύο περιπτώσεις δεν αναζήτησα τη διπλή αυτή ιδιότητα, το διπλό καπέλο και δεν το έχω φορέσει καν. Λοιπόν, πάρα πολύ γρήγορα να σας πω ότι υπήρχε καταρχάς θεωρήστε το διαφημιστικό διάλειμμα. Λοιπόν, μετά την εμπλοκή στι διαπραγματεύσει των κρατών μελών, η συμφωνία θα πρέπει να είναι ομόφωνη σε ό,τι αφορά το γενικό δίκαιο. Επανέρχεται στο Κοινοβούλιο αυτή η πρόταση στο πλαίσιο ενισχυμένη συνεργασία ε, που θα βοηθήσει, πιστεύω, να καταλήξει αίσιο πέρα. 18 κράτη-μέλη συγκεκριμένα ζήτησαν ε, η ενισχυμένη συνεργασία να εφαρμοστεί. Εδώ, Κύπρος τώρα ε, έχει και αυτή μπει σε αυτή την ενισχυμένη και άλλα πέντε κράτη το σκέφτονται. Οι τρει χώρε τη Βαλτική, η Ρουμανία και η Σλοβακία και ενδέχεται να προσχωρήσουν σε αυτή τη διαδικασία ενισχυμένη συνεργασία. Η πρόταση τώρα. Η πρόταση κανονισμού του 2016 και για τις δύο περιπτώσεις δεν είναι ταυτόσιμη με την πρόταση της Κομισιόν του 2011. Στι δύο προτάσει κανονισμού, λοιπόν, υπάρχουν διάφορε από τι ε, προτάσει που είχαμε εμεί διατυπώσει ω κοινοβούλε σε συζήτηση το 2013 και αντιστοιχούν στο κείμενο στο οποίο 23 κράτη-μέλη ε, θα έδιναν τη σύμφωνη γνώμη του στα τέλη του 2015. Αυτά για να δείτε έτσι λίγο και το συσχετισμό δυνάμεων. Πρόκειται για δύο κανονισμού πάρα πολύ χρήσιμου ε, για διεθνή ζευγάρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν είναι και λίγο όπω ξέρετε. Και δείχνουμε άλλωστε με αυτόν τον τρόπο ότι εν μέρει έχουμε αυτό το συγχρονισμό και τις επαφές διαφόρων εθνικοτήτων. Θέμα λοιπόν είναι η δικαιοδοσία, εφαρμοστέο δίκαιο, καθώς και αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων όταν υπάρχουν ε, συγκρούσεις ε, και έλλειψη συμβατότητας ε, κανόνων σε επίπεδο διαφορετικών κρατών μελών. Έχουν το πλεονέκτημα αυτοί οι κανονισμοί ότι ορίζουν με ξεκάθαρο τρόπο τη δικαιοδοσία που είναι αρμόδια να αποφαίνεται ε, για τα διάφορα αιτήματα όταν αυτά σχετίζονται ε, με την κληρονομική διαδοχή ενός συζύγου κλειπώντος ή ενός καταχωρημένου συντρόφου κλειπώντος και όταν υπάρχει αίτημα ε, αζυγίου, χωρισμού κτλ. Δεν επίπτει στο πεδίο του εδώ, στο πεδίο εφαρμογής μάλλον, η ικανότητα των συντρόφων, η ύπαρξη εγκυρότητα ή αναγνώριση ενός ε, γάμου ή μίας ε, συμβίωσης και το θέμα της διατροφής ε, και η κληρονομική διαδοχή ενός συντρόφου ή ενός σύζυγου που απεβίωσε να τα λέω όμως πιο αργά γιατί δεν θα καταλάβετε τίποτα μάλλον. Λοιπόν, η αρχή της επικουρικότητας σε θέμα οικογενειακού δικαίου διαφυλάσσεται 100%. Θέλω να κάνω μια διευκρίνηση τώρα στο πλαίσιο που ένα κράτος μέλος δεν αναγνωρίζει το γάμο ή την λόγο συμβίωση, καταλάβετε τι θέλω να πω, δίνεται η δυνατότητα στο δικαστήριο του ελόγου κράτους ε, να ε, θέσει την υπόθεση υπόψη ε, δικαστήριο μιας άλλης χώρας για να δοθεί από νομικής πλευράς μια σταθερή ε, σε ό,τι αφορά αυτή τη διαφορά Υπάρχει καθολική εφαρμογή, δηλαδή μπορεί να εφαρμοστεί και το δίκαιο ενός τρίτου κράτους. Ποια είναι η βασική βελτίωση με αυτό το κείμενο είναι ότι το εφαρμοστείο δίκαιο στα περιουσιακά στοιχεία του ζεύγους ισχύει για το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων που κατέχουν από κοινού. Όπου και αν είναι αυτά τα περιουσιακά στοιχεία Τώρα, για την εκτελεστότητα, την αναγνώριση των αποφάσεων κτλ. Το κείμενο, ω έχει αυτή τη στιγμή, εμπνέεται σε μεγάλο βαθμό από τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2013, ήδη το είπα αυτό. Άρα αναφέρει πολύ συγκεκριμένε διατάξει του κανονισμού για την κληρονομική διαδοχή, τη διασυνοριακή συγκεκριμένα κληρονομική διαδοχή. Αυτές οι δύο προτάσει κανονισμού συνιστούν πραγματική πρόοδο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τα διεθνή ε, ζευγάρια που είναι και το αντικείμενο αυτών των κανονισμών και που συχνά ε, αντιμετωπίζουν ενεκτήματα λόγω της έλλειψης σχετικής ε, νομοθεσίας. Μπορεί να υπάρχει σύγχυση, μπορεί να υπάρχει και αδικία, αλλά σίγουρα και ασάφεια δικαίου, κάτι που δυσκολεύει την επίλυση διαφορών στον τομέα αυτό. Θέλω να δώσουμε ως Κοινοβούλιο τη σύμφωνη γνώμη σε αυτές τους δύο ε, κανονισμούς ε, γιατί νομίζω ότι με την ε, από κοινού εξέταση των δύο εκθέσεων θα δώσουμε ικανοποίηση στα κράτη-μέλη που ήθελαν να υπάρξει μια παράλληλη διαδικασία. Σε επίπεδο Συμβουλίου κατέληξαν διαπραγματεύσει τελικά σε συμφωνία με βάση το πρώτο κείμενο και ζητεί το Συμβούλιο να ληφθούν υπόψη περισσότερες από τις προτάσεις του Κοινοβουλίου του 2013. Άρα νομίζω ότι μπορούμε να θεωρήσουμε ότι οι νέες προτάσεις συνιστούν θετικό συμβιβασμό που μας επιτρέπει να ρυθμίσουμε τις διαφορές και να προχωρήσουμε και εμείς και το Συμβούλιο. Άρα δεν θεωρώ σκόπιμο να προτείνω τροπολογίες. Γιατί θα μπορούσε αυτό να είναι αντιπαραγωγικό Μπορεί να μην ήθελα να το κάνω, αλλά σίγουρα θα δημιουργούσα δυσκολίες. Τρεις διευκρινήσει ακόμη, αν με επιτρέπετε. Πρώτα απ' όλα, να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι κάθε τροποποίηση θα έθετε υποφυσβήτηση το σέλ του, της συμφωνίας που επικυρώθηκε από τα κράτη-μέλη που συμμετέχουν στην ενισχυμένη συνεργασία και πρέπει να σας πω ότι οι διαπραγματεύσεις ήταν σκληρές, το γνωρίζετε, το φαντάζεστε. Άρα δεν θα ήθελα να καθυστερήσουμε. Είναι σημαντική η πρόοδος με αυτά τα ζευγάρια και γι' αυτό δεν πρέπει ε, να ε, παρανεγκρίνουμε αυτά τα δύο κείμενα πιστεύω. Διότι αλλιώς ε, δεν περιποιούμε κανένα αφού για αυτούς τους ανθρώπους. Τώρα τα... για τις προθεσμίες κατάστροπλα 4 Μαΐου. Άρα μπορούμε να συζητήσουμε τις τροπολογίες που ενδεχομένως κατατεθούν δεν είμαι υπέρ όπως ε, το καταλάβατε αυτό, στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Τελευταία πρόταση, τελευταία πληροφορία. Να εγκρίνουμε πριν τα τέλη Ιουνίου, αυτό θα ήταν ευκταίο. Και δεν νομίζω ότι είναι ανεύκτος ο στόχος, αλλά πολύ εφικτός αντίθετα. Και τέλος, αγαπητοί συνάδελφοι, αυτό το χρονοδιάγραμμα θεωρώ ότι είναι σημαντικό να το τηρήσουμε ώστε οι δύο εκθέσεις, τα δύο κείμενα αυτά, να εντριθούν από κοινού ταυτόχρονα σε επίπεδο Συμβουλίου τα κράτη-μέλη που συμμετέχουν στη διαδικασία ενισχυμένη συνεργασίας. Να έχουμε ολοκληρώσει δηλαδή παράλληλα αυτά τα δύο κείμενα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Και τώρα βάζω το άλλο μου καπέλο για να ακούσω τις παρεμβάσεις Ποιος θέλει το λόγο. Замбовски. Благодаря ви, уважаеми господин Кавада. Ευχαριστώ, κύριε Καβαντά. Αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα με την ευκαιρία να εκφράσω τις θέσεις μου για την έκθεση του κυρίου, για τις εκθέσεις του κυρίου Καβαντά σχέση με το εφαρμοστέο δίκαιο και την εκτέλεση αποφάσεων σχετικών με προβλήματα ζευγαριών. Άλλο βέβαια ο γάμος, άλλο τα καταχωρισμένα ζευγάρια και στο διεθνές δίκαιο ισχύει αυτό βεβαίως και ως προς τα περιουσιακά στοιχεία είναι δύσκολο να μιλούμε για ε, τα καταχωρισμένα ζευγάρια με όρους ε, παντρεμένων ζευγαριών. Αυτό διαφέρει από κράτος σε κράτος πάντα. Έχουμε δει εκθέσεις σε διαφορετικά ζητήματα, εκτελεστότητα αποφάσεων κτλ. Και αυτά δείχνουν ότι είναι διαφορετικοί οι δύο θεσμοί. Έτσι λοιπόν, διαρωτώ με τα κράτη-μέλη πώς μπορούν να δεχθούν αυτή την πρόταση, αφού είναι τόσο διαφορετική η κατάσταση σε χώρες ε, που δεν αναγνωρίζουν καν τα καταχωρισμένα ζευγάρια. Και άρα δεν έχουν εισαγάγει στο ιστορικό της δίκαιο αυτή τη σχέση. Γιατί θα πρέπει να αναγνωρίζουν οι χώρες αυτές θέματα περιουσιακών δικαιωμάτων και άλλα, τα οποία ρυθμίζει τη δικαιοδοσία άλλων κρατών, η νομιτάξη άλλων κρατών. Αν λοιπόν ε, δεν αναγνωρίζονται αυτές οι καταχωρισμένες ε, σχέσεις, τα καταχωρισμένα ζευγάρια, επιβάλλονται διακρίσεις που βέβαια δεν είναι προς όφελος των πολιτών. Και αυτό συνεπάγεται σοβαρές ε, συνέπειες στα κράτη-μέλη ως προς την υποχρέωση των κρατών μελών να αποδεχθούν τον κανονισμό και αμφιβολίες ως προς την αμφισβήτηση καλύτερα ως προς την αρχή της επικουρικότητας γιατί καλούνται τα κράτη να αναγνωρίσουν συνέπειες από τις καταχωρισμένες σχέσεις τα οποία, τα τις οποίες ε, τα ίδια δεν αναγνωρίζουν ως θεσμό στην ιστορική του ενόμη τάξη. Τον υποχρεωθούν λοιπόν τα κράτη να αναγνωρίσουν τα, τις συνέπειες ως προς την περιουσιακή κατάσταση. Φερρυπίν ε, αποφάσεις δικαστικές για την ε, κοινή περιουσία εμέσως αναγνωρίσουν αυτές τις ε, καταχωρισμένες σχέσεις αφού αναγνωρίζουν τις συνοηπιές τους, όπως αναφέρεται στο κείμενο. Η Επιτροπή δεν προτείνει εκτίμηση των συνεπειών της προτινόμενης πρότασης κανονισμού. Η Επιτροπή μας λέει ότι θα ακολουθήσει αξιολόγηση συνεπειών για την κάθε πρόταση. Δύο εκατομμύρια είναι τα διεθνή ζευγάρια που έχουν εγκατασταθεί σε διαφορετικές περιοχές, αλλά για τα καταχωρισμένα ζευγάρια πάλι η κατάσταση θα πρέπει να είναι διαφορετική και δεν είναι δυνατόν να υποχρεωθούν τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν αυτόν τον κανονισμό, γιατί αυτός δεν πρέπει να είναι εφαρμόσιμος όταν σε κάποια κράτη δεν γνωρίζονται τα καταχωρισμένα ζευγάρια και έτσι θα έχουμε πολλές περιπτώσεις άνθρωπων οι οποίοι δεν θα μπορούν να έχουν την απόλαυση των δικαιωμάτων τους. Ερωτώ λοιπόν γιατί να μην είναι πιο ευέλικτη η πρόταση, να μην αφήνει περιθώριο ε, διακριτικής ευχαίριας προς τα κράτη-μέλη. Μια ευελιξία που θα αποτελούσε άλλωστε και την ουσία αυτής της ενισχυμένης συνεργασίας τα 20 τελευταία έτη. Οι εθνικές νομοθεσίες έχουν ε, ρυθμίσει διαφορετικά τις καταστάσεις. Τα καταχωρισμένα ζευγάρια αναγνωρίζονται σε ορισμένες ένομες τάξεις και έτσι ώστε έπρεπε να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να διευκολύνουμε βεβαίως την κινητικότητα των ανθρώπων και την αξιοποίηση ρυθμίσεων κοινών προς τα κράτη-μέλη χωρίς ωστόσο να ε, περιστέλουμε τις δυνατότητες ένα κράτος μέλος να επιβάλλει ένα διαφορετικό καθεστώς στην εσωτερική του ένωμη. Εντάξει, ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ κύριε Τζαμπάσκι, κύριος Φως. Κύριε Φως, Πρόεδρε, θυμάμαι ακόμη τότε που εκείνο το θέμα που μας ανέφερε τώρα ο κύριος Τζαμπάσκι, τρία-τέσσερα χρόνια, ε, ήγηρε πολλές ανησυχίες, ευαισθησίες και αντιδράσεις, αλλά θα ήθελα να συμφωνήσω με την πρότασή σας εγώ και να υποστηρίξω το κείμενο όπως το έχετε καταθέσει. Είναι σημαντικό, πιστεύω, με την ευκαιρία αυτή να προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατό σε μια συμφωνία γιατί έχουμε να κάνουμε με αίτημα του Κοινοβουλίου του 2013 ήδη, το οποίο σε μεγάλο βαθμό έχει γίνει δεκτό, έχει συμπεριληφθεί στο τωρινό κείμενο και βλέπω ότι ε, οδηγούμαστε σε καλά συγκεκριμένα και ε, σημαντικά αποτελέσματα εφόσον αυτή η διαδικασία ολοκληρωθεί επιτυχώς. Είναι ε, ισορροπημένες οι προτάσεις ιδιαίτερα για τα καταχωρισμένα ζευγάρια, τα κράτη εκείνα συγκεκριμένα τα οποία δεν έχουν εισαγάγει αυτό το σύστημα στην ε, εσωτερική του ένωμη τάξη δεν υποχρεούνται να την εισαγάγουν, να εισαγάγουν το θεσμό αυτό από την πίσω πόρτα. Το είχαμε ξανασυστήσει και πιο, πριν δύο-τρία χρόνια. Δεν θα πρέπει να υποχρεωθούν στην εισαγωγή ενός νέου θεσμού ε, εμέσως. Υπάρχουν κάποιες αιτιολογικές σκέψεις τελευταία ανάλυση και άρθρα της πρότασης που αναφέρουν συγκεκριμένα ότι το ζήτημα των καταχωρισμένων ζευγαριών ισχύει μόνο για τις χώρες που αναγνωρίζουν, ωστόσο οι υλικέ και περιουσιακές συνέπειες δεν μπορούν να αναπτυχθούν ε, πέραν ε, του απλού ζητήματος αυτού του περιουσιακού, δηλαδή δεν μπορούν να επηρεάσουν την ουσία, το βασικό ζήτημα της αναγνώρισης του καταχωρισμένου ζευγαριού, δηλαδή δεν μπορεί να γίνει επέμβαση στην εσωτερική ένωση τάξη, δεν παρεμβαίνουμε στο εθνικό δίκαιο, τα κράτη-μέλη ε, διατηρούν την ε, δυνατότητα να αποφασίσουν τα ίδια εάν θέλουν να ρυθμίσουν στο εσωτερικό τους δίκαιο ε, το θεσμό του καταχωρισμένου ζευγαριού ή όχι. Έτσι λοιπόν, είτε πρόκειται για ζευγάρια με γάμο ή καταχωρισμένα μόνο, ε, δεδομένου ότι είναι όλο και μεγαλύτερος ο αριθμός εκείνων που έχουν διεθνή χαρακτηριστικά και άρα κινούνται περισσότερο από τη μία χώρα στην άλλη, είναι σημαντικό να προχωρήσουμε στη ρύθμιση των εκκρεμών ζητημάτων σε σχέση με την περιουσία των συζύγων και τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία όταν πρόκειται για τα καταχωρισμένα ζευγάρια βεβαίω. Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, το κληρονομικό δίκαιο έχει ήδη ρύθμιση σε υπερσυνοριακό επίπεδο και γι' αυτό θεωρώ ότι υπάρχει ανάγκη και στην περίπτωση των ε, περιουσιακών στοιχείων των ε, ε, ζευγαριών να υπάρξει σχετική ρύθμιση. Το ταχύτερο δυνατό θα σημειώσω πρέπει να προχωρήσουμε σε μία ρύθμιση. Ε, και στις δύο περιπτώσεις των, κυμα... κειμένων έχουμε να κάνουμε με ενισχυμένη συνεργασία και με τα κράτη-μέλη και αυτό υπογραμμίσω και πάλι καθώς το κείμενο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2013 βλέπουμε να αντικατοπτρίσει στο κείμενο που έχουμε μπροστά μας δεν έχω ε, επιφυλάξει ως προς την ουσία της υπόθεσης και διαδικαστικά θα θεωρούσα πολύ εύστοχο εάν μπορούσαμε να εγκρίνουμε τα δύο κείμενα μαζί και γρήγορα. Ευχαριστώ. Κυρία Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με πάσα ειλικρίνεια λέω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε σήμερα το σύνολο αυτό μέτρων. Το 2013 ήμουν και εγώ εδώ και μάλιστα ω εισηγήτρια τη Επιτροπή των Πολιτικών Ελευθεριών είχα αναλάβει την επεξεργασία του θέματο. Θυμάμαι πολύ καλά όλη τη συζήτηση και πόση απογοήτευση αισθανόμουν κάθε φορά που έβλεπα ότι δεν προχωρά η υπόθεση για τα κράτη-μέλη δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν απλά και μόνο και με βάση βέβαια αυτή την αρχή της ομοφωνίας με αυτά τα προβλήματα. Είναι πολλά τα ζευγάρια με διεθνή χαρακτήρα, με διαφορετικές εθνικότητες που περνούν μέσα από τα πάθη του Ιώβ για να μπορέσουν να ρυθμίσουν τα ζητήματά τους και βέβαια και τα ε, περιουσιακά. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάντοτε θεωρούσε σημαντικό και το υπογράμμισε τα δύο κείμενα αυτά, κληρονομικά δηλαδή και περιουσιακά συζύγων, να ρυθμιστούν ταυτόχρονα γιατί ήταν για πολλά κράτη-μέλη, όχι για όλα, πάρα πολύ σημαντικό ε, τόσο για τα ζευγάρια με γάμο όσο και τα καταχωρισμένα ζευγάρια να υπάρχει η ταυτόχρονη ρύθμιση των ζητημάτων. Βεβαίω, σεβόμαστε το γεγονό ότι σε ορισμένα κράτη-μέλη, και το έχουμε πει ανέκαθεν αυτό, δεν αναγνωρίζονται τα καταχωρισμένα ζευγάρια. Γι' αυτό και πάντοτε υπογραμμίζαμε ότι το σεβόμεθα, ότι δεν θα υπογραφεί κανένα κράτο να ρυθμίσει κάτι το οποίο δεν επιθυμεί να ρυθμίσει. Ούτω ή άλλω, δυνάμει και των συνθηκών τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουμε κανένα τέτοιο δικαίωμα ή αρμοδιότητα για το άρθρο 9 παράγραφος 1 του κανονισμού για, τα κατοχωρισμένα ζευγάρια. Ξεκάθαρα αναφέρεται ότι μπορούν να δηλώσουν τα δικαστήρια ε, να ε, δηλώσουν ότι είναι αναρμόδια τα ίδια σε περίπτωση που το εθνικό δίκαιο δεν αναγνωρίζει τα κατοχωρισμένα ζευγάρια. Κανένα κράτος λοιπόν και κανένα δικαστήριο δεν υποχρεούται να λάβει αποφάσεις οι οποίες θα αντέβαιναν στην εσωτερική ένωμη τάξη του κράτους. Απλώς θέλουμε να υπάρχει η δυνατότητα. Αυτό ε, επιδιώκουμε και σε αυτό συμμερίζομαι και την άποψη του εισηγητού ότι πρέπει να προχωρήσουμε ταχύτατα από το 2011 έχουμε αρχίσει να επεξεργαζόμαστε αυτές τις προτάσεις και θα σας πω το εξής. Εγώ δεν είμαι καθόλου υποστήρικτρια της ενισχυμένης συνεργασίας γιατί γίνεται μόνο γνωμοδότης από το Κοινοβούλιο, έχει συμβουλευτικό μόνο ρόλο και μετά δεν μπορεί να παρέμβει άλλο. Αλλά από όσα είχε αποφασίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2013 όλες οι προτάσεις έχουν γίνει δεκτές. Αυτό λοιπόν είναι τεράστια ευκαιρία, έστω και αν δεν θέλαμε να προχωρήσει έτσι, αν θέλαμε άλλη διαδικασία, τώρα έχουμε αυτό που επιδιώκαμε και πρέπει να δεχθούμε τον κανονισμό όπως έχει και πιστεύω ότι στην ομάδα μου δεν θα προκύψει καμία τροπολογία, διότι θέλουμε να διασφαλίσουμε πώς το δίκαιο αυτό και το δικαίωμα αυτό θα εγκαθιδρυθεί για τους πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό, το οφείλουμε στους πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυριολεκτικά το λέω, και πάνω απ' όλα απευθύνω έκκληση στα κράτη-μέλη, εκείνα τα οποία ακόμη δεν έχουν ε, συμπράξει, να συμπράξουν γιατί αφορά η ρύθμιση αυτή πάρα πολλούς ανθρώπους και πρέπει να τους βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς να βρουν την ασφάλεια δικαίου, τη ρύθμιση αυτή που σήμερα δεν υπάρχει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το Συμβούλιο, κυρία Κέντα μου. Καλημέρα κύριε Καβαντά. Σας ευχαριστούμε, σας ευχαριστούμε που δίνετε το λόγο στην ε, Ολλανδική Προεδρία. Σας ε, επιβεβαιώνω ότι για μας το θέμα αυτό είναι μεγάλης προτεραιότητας. Ο κανονισμός είναι πολύ σημαντικός για τα μεικτά ζευγάρια και ξέρουμε όλοι ότι υπάρχει μακρά ιστορία σε αυτό το θέμα. Γι' αυτό η Προεδρία έχει τη φιλοδοξία να υιοθετήσει τις προτάσεις πριν από την 1η Ιουλίου. Για να προχωρήσουν οι εργασίες πιο γρήγορα στο Συμβούλιο, ε, πολιτική πολιτικής σημασίας, η Προεδρία αποφάσισε να αντιμετωπίσει τις τρεις προτάσεις ε, σε μεγάλο βαθμό ταυτόχρονα. Δηλαδή την πρόταση για την απόφαση έγκρισης από τη μία και τις δύο προτάσεις για τους καουνισμούς Απ' την άλλη, αυτό γίνεται χάρη στο ότι η Κομισιόν δημοσίευσε τις τρεις προτάσεις την ίδια μέρα, αρχές Μαρτίου δηλαδή. Σε ό,τι αφορά τις εργασίες του εσωτερικού του Συμβουλίου, Συμφωνώ μαζί σας ότι μόνο κάποιες λίγες τεχνικές τροποποίησεις έχουμε εισαγάγει για να διευκρινίσουμε κάποια στοιχεία που συνδέονται με το γεγονός ότι τώρα χρησιμοποιούμε το εργαλείο της ενισχυμένης συνεργασίας. Ο πυρήνα των κειμένων δεν έχει αλλάξει, το τονίζω. Επίσης έχω και άλλα καλά νέα, φρεσκότατα από το Συμβούλιο, δηλαδή σήμερα το πρωί το θέμα αυτό εξετάστηκε το Κορεπέρ και συμφώνησε το Κορεπέρ και για τις τρεις προτάσεις ταυτόχρονα. Μια και συμφώνησε τώρα το Κορεπέρ των κειμένων, η Προεδρία σκοπεύει να στείλει την πρόταση για απόφαση έγκρισης στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της 12ης Μαΐου, ούτως ώστε να υπάρξει έγκριση και από το Κοινοβούλιο για την απόφαση. Εννοείται ότι θα περιμένουμε με ενδιαφέρον την έγκρισή σας. Σε ό,τι αφορά τις προτάσεις για τους κανονισμούς, θα σταλούν στο Συμβούλιο Τζάι ε, της 9ης ε, Ιουνίου για τη γενική προσέγγιση και θα περιμένουμε επίσης με ενδιαφέρον την άποψη του Κοινοβουλίου για τους δύο κανονισμούς. Ελπίζουμε ότι μπορούμε να βασιστούμε στην ε, στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αυτά τα σημαντικά θέματα για τους πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης και σας ευχαριστούμε ήδη για την καλή συνεργασία μέχρι τώρα. Ευχαριστούμε για τα φρέσκα νέα, κυρίως. Νομίζω ότι διευκολύνεται τις εργασίες μου. Ε, για τις τροπολογίες έχουμε προθεσμία μέχρι τις 3 Μαΐου. Πάμε στο σημείο 12 και κλεισμένο των θυρών θα γίνει αυτό. Όλοι όσοι δεν έχουν θέση εδώ παρακαλώ να εγκαταλείψουν την αίθουσα. Δύο λεφτά διάλειμμα γιατί θα βγείτε τρέχοντας.